Τελειώσαμε με αυτό το σημείο και αύριο στις 11.30 θα ψηφίσουμε το σχετικό ψήφισμα. Πάμε τώρα στις τοποθετήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 150. Είναι οι τοποθετήσεις ενός λεπτού και θα έχουν την προτίμηση οι βουλευτές που βάσει του άρθρου 150 στην προηγούμενη Ολομέλεια δεν πήραν το λόγο. Θα προηγηθούν λοιπόν αυτό που μίλησαν ήδη. Ο κύριος Ογκουρεάνου λοιπόν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, στις 4 Φεβρουαρίου του 2010 ο Ρουμανός, Ρουμάνος Πρόεδρος να εκείνωσε την συμμετοχή της Ρουμανίας σε το ο αντιπυραυλικό σύστημα ε, και αυτό, του ΝΑΤΟ και αυτό πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται για ένα σύστημα ε, εναντίον της Ρωσίας. Είμαστε ε, ένας τέρος των άλλων κρατών και θα υπάρξει μία συμφωνία η οποία θα μπορέσει μπορέσει να ενισχύσει τη θέση των Ευρωπαίων ε, εταίρων και ελπίζω ότι θα υπερψηφιστεί αυτή η σημαντική συμφωνία. Για ένα λεπτό η κυρία Δαντσίλα. Elle n'est pas là Elle n'est pas présente δεν είναι εδώ. Η κυρία Σκριζντιλεύσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για την κατάσταση των ε, συμπολιτών μου στη Λιθουανία όπου τα ουσιαστικά τα δικαιώματα των, ε, της, της πολωνικής μειονότητας καταπατούνται ε, παρόλο που αποτελούν ένα μέρος του πλήθη δεν μπορούν να εξασκήσουν την ε, μητρική τους ε, γλώσσα τα πολωνικά ονόματα ε, προσαρμόζονται στην λιθουανική μορφή και ε, υπάρχει ε, μία, ε, μία διάκριση εναντίον τους. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε αν μπορούμε να ζήσουμε σε μία Ευρώπη ψευδεστήσεων ή πραγματικών αξιών. Εάν θα δεχθούμε αυτή την καταπάτηση των δικαιωμάτων ή θα θέλουμε να οικοδομήσουμε μία Ευρώπη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Περιγιού. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ανακοινώσω κάτι. Ότι στη Βαλένσια υπάρχει μια παραλιακή συνοικία ιστορική, τον Παρανιάλ, που θα καταστραφεί σύμφωνα με το νέο σχέδιο, πολυδομικό σχέδιο. Ξεσηκώθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι, προσέφυγαν στο δικαστήριο και το δικαστήριο αποφάσισε να σταματήσουν τα έργα. Οι αρχές όμως αποφάσισαν με διοικητικά μέτρα να προχωρήσουν. Ζητώ λοιπόν να υποστηριχθεί η γειτονιά του Καμπανιάλ στη Βαλένσια από την καταστροφή. Ο κύριος Μπουσόη, για ένα λεπτό. Έλαβα μέρος στην ομάδα κοινοβουλευτικής συνεργασίας Ένωσης Μολδαβίας ήταν ενθαρρυντική για τις διμερείς μας σχέσεις και για την βελτίωση των σχέσεων Μολδαβίας με Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν σημαντικές πρόοδοι και αυτή η πρόοδοι είναι σημαντικό σημάδι για την βούληση της Μολδαβίας να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περασμένη εβδομάδα συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση της κυβέρνησης εκεί για μεταρρυθμίσεις και εκδημοκρατισμό. Χαιρετίζουμε τη νέα συμφωνία σύνδεσης που ξεκίνησε να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζει την υποστήριξη αυτή τη συμφωνία και να προχωρήσει σε συμφωνία ελεύθερη θεωρήσεων το Κοινοβούλιο και η Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει την κυβέρνηση αυτή με οικονομική βοήθεια που θα πρέπει να χορηγηθεί το ταχύτερο δυνατόν και με την εμπειρογνωμοσύνη των, της Ένωσης για μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και στην οικονομία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαρνέκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δυστυχώς πρέπει και πάλι να επανέλθω εις ε, την κατάσταση ε, της πολωνικής μειονότητας στη Λιθουανία, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κανονικά θα έπρεπε να ε, γίνονται σεβαστές όλες οι ε, ε, αρχές της Ευρώπης σε όλες τις χώρες αλλά εδώ βλέπουμε ότι η πολωνική μειονότητα αποτελούν, αποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσμού έχουμε όμως πρόβλημα με τα σχολεία με το θέμα της εκπαίδευσης και προβλέπεται να μειωθούν και να συρρυκνωθούν οι ε, τάξεις ε, στα σχολεία ε, και αυτό είναι μία ασυμμετρία διότι η λιθουανική μειονότητα στην Πολωνία χαίρει κάθε εκτιμήσεως και έχει όλες τις δυνατότητες. Θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Για ένα λεπτό ο κύριος Μπάτερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πήγα σε μια δεξίωση για το Shenyong Performing Group. Πέρυσι είχα την ευκαιρία στο Λονδίνο να δω την παράσταση τους και σκοπός τους είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον και να δείξουν την παραδοσιακή κινέζικη κουλτούρα που βεβαίω μια κουλτούρα που η κινέζικη κομμουνιστική κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να καταστρέψει μέχρι τώρα. Με λίγο μου έμαθα μέχρι σήμερα το βράδυ ότι μια παράστασή τους την, τον Απρίλιο στη Ρουμανία ακυρώθηκε μετά από πίεση της κινέζικης κυβέρνησης. Είναι παράδεκτο η Ρουμανία που λέει ότι είναι δημοκρατική επιτρέπεται να δεχτεί πιέσεις τέτοιες από μια κομμουνιστική τυραννία. Θα, να σας πω επίσης ότι η Σενγιόν δημιουργήθηκε επίσης και την φιλοσοφία για την ε, ανοχή και Γι' αυτό λοιπόν και τους φοβούνται ε, στην κομμουνιστική κυβέρνηση του Πεκίνου. Θα ήθελα πάντως να προτείνω στον πρόεδρο κύριο Μπούζακ να καλέσουμε το Σεν για να μας κάνουν μια παράσταση εδώ στο Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατόν και αυτό θα είναι σαφές κίνηση, σαφής κίνηση υποστήριξης σε αυτούς τους ε, ε, δημοκρατικούς αγωνιστές κατά της κινητικής κυβέρνησης. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με την ευκαιρία αυτή να καταδικάσω την, πλαστή, την παράνομη χρήση των ευρωπαϊκών διαβατηρίων της Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιρλανδίας στην δολοφονία αυτή στο Ντουμπάι. Η αστυνομία της Ντουμπάι είναι σίγουρη σχεδόν ότι οι Ισραηλινοί ε, διέπραξαν το έγκλημα χρησιμοποίησαν πλαστιγραφημένα βρετανικά διαβατήρια για την διαπράξη εγκλήματος σε τρίτη χώρα. Αυτό είναι καταπαράβαση κατά παράβαση της νομοθεσίας μας και εμείς πάντα ήμασταν ειρηνικοί και επιτρέπεται να ταξιδέψουν οι πολίτες μας σε μέρη που συχνά απαγορεύεται. Αυτό διακυβεύει τη θέση μας αυτή και καλό την τη εκπρόσωπο ιδιαίτερα να διαρευνήσει το θέμα και εάν η, η κυβέρνηση της Μοσάντ κρύβεται πίσω από όλα αυτά, τότε να δοθεί ε, αποζημίωση σε εμάς και στις άλλες χώρες που συμμετείχαν. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο για ένα λεπτό, αλλά δεν είναι ο ίδιος κύριος Κέλλη, είναι ο κύριος Άλαν Κέλλη. Κάποια στιγμή θα ξεκαθαρίσουμε το θέμα. <coughs> το θέμα των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να αναθεωρηθεί διότι στην προηγούμενη θητεία της Επιτροπής βασίστηκε ε, κανείς στις ε, τότε ισχύουσες στατιστικές του Ευρωστάτ ενώ τώρα πρέπει κανείς να ε, διαπιστώσει ότι η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά. Εάν κοιτάξει κανείς τη δικιά μου χώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μία σημαντική αύξηση ε, των ε, προβλημάτων στο Λίμερικ σε πολλές ε, περιοχές όπου έχει αυξηθεί η ανεργία και υπάρχει επιδότηση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά οι στατιστικές του 2007-2008 είναι αναχρονιστικές. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την οικονομική εξέλιξη και να μην παραμένει σταθερή στις θέσεις της. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τούρκ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο αγαθό που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο είναι το σκυλί Υπήρχε ε, ε, μία περίπτωση στη Γαλλική Επανάσταση, μία ευγενής η οποία είχε πει ότι τελευταίως αρχίζω να συμπαθώ περισσότερο τα σκυλιά από τους ανθρώπους και ε, έχουμε όμως πάρα πολλούς λάτρεις των σκυλιών στη χώρα μου οι οποίοι ενοχλούνται ε, για τον αριθμό των ε, ε, σκυλιών που σκοτώνονται σε τροχαία ατυχήματα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μία νομοθεσία από το Κοινοβούλιο η οποία όμως προβλέπει ότι θα σκοτώνονται τα αδέσποτα ενώ όμως εφόσον έχουμε σκυλιά δεν έχουμε φίδια και ε, ε, διάφορα άλλα ζώα. Οπότε δεν ε, πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε στην τρίτη χιλιετηρία και ο άνθρωπος αγαπάει και τον άνθρωπο και τα ζώα. Συνάδελφοι, καταγγείλω την κατάσταση για τον χείριο τομέα στην Καταλωνία. Μειώνονται οι τιμές εδώ και ένα χρόνια και για πολλούς μήνες είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Ένας από τους λόγους για το οποίο συμβαίνει αυτό είναι από τις εισαγωγές χείριου κρέατος από τις αναδιόμενες χώρες. Πολλές φορές αυτές οι εισαγωγές δεν ελέγχονται επαρκώς στα ευρωπαϊκά τελωνία. Σε πολλές περιπτώσεις αυτά, αυτές οι εισαγωγές χείριου κρέατος πληρούν πολλές οδηγίες που απαιτούνται και φαίνεται ότι το ίδιο θα συμβεί και τα επόμενα χρόνια. Οι όλο και μεγαλόμενες αυξανόμενες απαιτήσει από τους Ευρωπαίους παραγωγούς αλλά κανένας έλεγχος για τις εισαγωγές. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι σαφής περίπτωση αθέμη του ανταγωνισμού. Έτσι η Ευρώπη θα χάσει τους παραγωγούς χειρίου κρέατος και τους γεωργούς του και χωρίς αυτούς η Ευρώπη θα χάσει ένα σημαντικό τμήμα του γεωργικού της τομέα. Αυτές τις ανησυχίες ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ευχαριστούμε κύριε Τρεμόσα. Για ένα λεπτό, ο κύριος Τομασεύσκη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να επανέλθω στο θέμα της πολωνικής μειονότητος στη Λιθουανία, διότι τα δικαιώματα της ε, μειονότητος περιορίζονται. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές όπου υπάρχει απαγόρευση να χρησιμοποιούνται οι πινακίδες και στις δύο γλώσσες, ενώ υπήρχαν επί 20 χρόνια. Υπάρχουν προβλήματα με τα σχολεία. Όσον αφορά ε, τα ε, δημόσια έγγραφα, τις ταυτότητες και τα διαβατήρια δεν χρησιμοποιείται πλέον η πολωνική γραφή, ε, δεν επιστρέφονται οι περιουσίες και το σύνολο βίλια έχει φαρπαγεί από το κράτος. Τα δικαιώματα λοιπόν της μειονότητας αυτής θα πρέπει να γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τις αρχές της ποικιλομορφία. Ευχαριστώ κύριε Τομασεύσκη. Η κυρία Μαγκίνες για ένα λεπτό. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε στην γεωργική παραγωγή χαμηλού κόστους και μένα με ανησυχεί το θέμα αυτό. Όμως ανησυχώ περισσότερο για την Κομισιόν και το πώς αυτοί βλέπουν τη γεωργική παραγωγή, γιατί στη στρατηγική του 2020 φαίνεται ότι σχεδόν έχουν ξεχάσει αυτό το ζωτική σημασία τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό την Κομισιόν να μην αγνοήσει αυτή τη σημαντικό τομέα και ελπίζω να μην θεωρείται ότι δεν είναι πλέον σημαντικός μια και τώρα θα μεταρρυθμίσουμε και τον υπολογισμό της Ένωσης. Υπενθυμίζω στην Κομισιόν ότι γεωργικό ε, διατροφικός τομέας είναι σημαντικός για λόγους υγείας, διατροφής και θέσης απασχόλησης στην Ήπεθρο και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στρατηγική το 2020 και χαιρετίζω και τις οργανώσεις γεωργών στην Ιρλανδία που εκπροσωπούν άνδρες και γυναίκες και τους ευχαριστώ που μου σημείωσαν το θέμα αυτό. Η κυρία Τικάου για ένα λεπτό. Muchas gracias, señor presidente. La începutul anului rata șomajului în zona euro era de 10%. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανεργία στην Ένωση στην αρχή του έτους ήταν 10% για τους νέους η ανεργία είναι 21%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περίπου 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις και το 99% αυτών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 2 τρίτα του εργατικού δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα απασχολείται από ΜΜΕ. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να προωθήσει ένα πακέτο για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να υπερνικήσουν την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Θα πρέπει να είναι πιο εύκολο να συστήσει κανένας μια ΜΜΕ και τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση και το 7ο ερευνητικό πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο να μπορέσουν δηλαδή τα ΜΜΕ, οι ΜΜΕ να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και όπως σημαίνει και με τους γεωργού θα πρέπει να υπάρχουν κρατικές εγγυήσει για δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να υπερνικήσουν την κρίση. Ευχαριστώ κύριε Τικάου. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Πρόεδρε, το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης στην ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονο σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή ένωση αυτό είναι γνωστό και οι λόγοι είναι ποικίλοι από τη γεωγραφική της θέση μέχρι και τη μεγάλη έκταση των θαλάσσιων συνόρων της. κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι τουλάχιστον πρόχειρη η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης αυτή την περίοδο για την χωρίς προηγούμενο διευκόλυνση της απόδοσης ελληνικής ηθαγένειας στους μετανάστες και εμφανίζεται το παράδοξο η πρόταση της κυβέρνησης της χώρας με το πιο έντονο πρόβλημα να περιλαμβάνει τις πιο επίοικείς ρυθμίσεις σε κάθε επίπεδο σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνει αντί να αποθαρρύνει τη λαθρομετανάστευση σε βάρος της νόμιμης μετανάστευσης υπονομεύει την κοινωνική ε, συνοχή αντιμετωπίζει αποσπασματικά το θέμα εξετάζοντας αποκλειστικά τον τελευταίο κρίκο μιας αλυσίδας περιλαμβάνει την παράνομο είσοδο στη χώρα το άσυλο την απέλαση την άδεια παραμονής και εργασίας στην ευρωπαϊκή ένωση και ανοίγει το παράθυρο για την απόκτηση ευρωπαϊκής ηθαγένειας σε απροσδιόριστο αριθμό λαθρομεταναστών. από την ε, οπτική αυτή γωνία είναι ένα ζήτημα ευρωπαϊκό που θα πρέπει να μας απασχολήσει έντονα το προσεχές διάστημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Ο κύριος Ενθιού για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο σεβασμός ιδιωτικής ζωής είναι ένα νέο θέμα, ιδίως γιατί έχουμε νέες ηλεκτρονικές τεχνολογίες οι οποίες είναι προς όφελος των ανθρώπων σε πολλούς τομείς αλλά υπάρχει μία έλλειψη ε, αξιοπιστίας και ε, σεβασμού των προσωπικών δεδομένων. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορεί ο κάθε πολίτης να παρακολουθεί και να ελέγχει ε, την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του. Δεν μπορεί η προστασία αυτή να επιλύσει όλα τα προβλήματα και τον τελευταίο καιρό έχουμε λάβει στοιχεία τα οποία μας προτρίνουν να προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή. Θεωρούμε όμως ότι είναι ακόμη ανεπαρκή σε πολλούς τομείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Βλάσεκ, για ένα λεπτό. Εδώ και έξι μήνες ο Καναδάς επανέφερε την απέτηση θεώρησης για τους πολίτες της Τσεχίας και ο λόγος για τον οποίο το έκαναν αυτό είναι διότι οι Ρώμα ζήτησαν, ζητούσαν άσυλο στον Καναδά. Πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μας έχουμε τις ίδιες συνθήκες για όλους, είτε είναι Τσέχοι, Σλοβάκοι, Βιετναμέζοι ή Ουκρανοί ή ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη φυλή. Η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δηλώνει ότι όλοι έχουν ισότιμα δικαιώματα. Η δικαιολογία του Καναδά είναι η Ρώμα. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι εξαιτία μίας μόνο ομάδας άλλαξαν τις προϋποθέσεις για όλους και θα πρέπει να ανακληθεί αυτή η απέτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δίας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις 11 του μηνός είπε όχι το σώμα στο SWIFT, στο πρόγραμμα παρακολούθησης δηλαδή των συναλλαγών της τρομοκρατίας. Τώρα όμως η Κομισιόν έχει μία νέα εντολή για το θέμα. Ρωτώ λοιπόν το Προεδρείο του Κοινοβουλίου, όχι εσάς, τον Πρόεδρο. Ρωτώ, οι Ηνωμένε Πολιτείε μετά από όλη αυτή την αποτυχία θεωρούν συνομιλητή τους την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διαπραγματεύονται διμερός. Αν συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη, ζητώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη θέση του στη διαπραγμάτευση αυτή. Ο κύριος Μποργέτσο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις 23 Φεβρουαρίου ρήπαν σημαδεύτηκε από τη ρήπανση του Λάμπρου, ενός παραποτάμου του Πο, του Πάδου, λόγω των διαρροών ε, ενός εγκατελελειμμένου δηληστηρίου. Η ρήπανση λοιπόν του πάδου μπορεί να οδηγήσει στην ρήπανση όλες τις κοιλάδας της Λομβαρδίας και της Αδριατικής. Ζητούμε λοιπόν να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει το περιβάλλον στις περιοχές της κοιλάδας του Πάδου αλλά να παρέμβει και για την αποκατάσταση της περιοχής που έχει πληγεί από την οικολογική καταστροφή. Κυρία Καρβάλο, ναι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι περιφερειακές διαφορές είναι μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο η πολιτική συνοχής να υποστηρίξει τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και χαίρομαι για την πρωτοβουλία για την Βαλτική θάλασσα και για την στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη. Έτσι έχουμε μια διαδικασία προβληματισμού για τη δυνατότητα νέων στρατηγικών στρατηγιών και για άλλες περιφέρειες. Στην νοτιοδυτική ε, περιοχή της Ευρώπης ή στις, ε, στα Κανάρια και στην Μαδέιρα που έχουν κοινέ προκλήσεις και μια στρατηγική για αυτήν την περιοχή θα βελτιώσει τα μέσα επικοινωνίας, το περιβάλλον, την επιστημονική ανταλλαγή δεδομένων και θα διευκολύνει την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Θα είναι επίσης και μια ανάπτυξη της Ευρώπης προς τον Ατλαντικό και θα είναι άλλη μια γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική. Ευχαριστώ κύριε Καρβάλιο. Ο κύριος Άλβες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τις νησογειωτικές περιοχές οι αερομεταφορές είναι το μόνο μέσο μεταφοράς και για τους επιβάτες και για το φορτίο υπάρχουν πολλές νησιωτικές περιοχές όπου είναι δύσκολες οι αερομεταφορές και υπάρχουν περιοχές όπου οι αζόρες και δεν, οι οποίες δεν είναι ελκυστικές για τις εμπορικές εταιρείες. Κατά συνέπεια η τιμή των εισιτηρίων είναι πολύ ακριβή, είναι εις βάρος της κινητικότητα του πληθυσμού και των τουρισμού και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα δυσμενές για μια τέτοια εποχή κρίσης που διανύουμε. Χρειάζεται λοιπόν προσωρινή υποστήριξη έτσι ώστε και να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η αγορά και να μπορέσουν και αυτές οι περιοχές με μεγάλο τουριστικό δυναμικό να επωφεληθούν από τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ο κύριος Σικέρσκι για ένα λεπτό.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 έχουν διακηρύξει το τέλος της οικονομικής κρίσης αλλά δεν μας δίνουν τα στοιχεία, τα στοιχεία για την ανεργία τα οποία είναι ανησυχητικά. Έχουμε πέραν των 23 ε, εκατομμυρίων ε, ε, ανέργων στην Ευρώπη πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και η κατάσταση των νέων ανέργων είναι επίσης πολύ ανησυχητική στους πέντε νέους στην Ευρώπη είναι άνεργος και αυτό θα έχει κοινωνικές επιπτώσεις όπως τα ναρκωτικά, ο αλκοολισμός, παθολογίες και εγκληματικότητα. Όσον αφορά τις διεξόδους για το μέλλον θα πρέπει να ενισχύσουμε την εσωτερική μας αγορά. Δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τις δυνατότητες του εσωτερικού ευρωπαϊκού χώρου θα πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική οικονομική ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θανασέσκου για ένα λεπτό. Din cauza expirării standardului de bune practici de... Πρόεδρε, στις αρχές Φεβρουαρίου το Εθνικό Ινστιτούτο της Βουκουρεστίου για την μικροβιολογική ανάπτυξη δεν έχει πλέον άδεια για την κατασκευή και θέση εμπορία σε αγορά των εμβολίων εξαιτία της περάτωσης της άδειά τους. Τα μέτρα αυτά εγκρίθηκαν από την διοίκηση του Ινστιτούτου και αναμένουμε ότι στα μέσα Απριλίου θα ξαναανακτήσει την άδεια αυτή. Αυτή η αναστολή για μερικούς μήνες ενός τέτοιου σημαντικού Ινστιτούτου είναι πολύ επικίνδυνο γεγονός. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ελέγχουν τακτικότερα τέτοιου είδους καταστάσεις για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ανακλήσεις των αδειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρασε η μισή ώρα. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης. Όπου τρέφω στο πρόσωπό σας υποβάλλω το αίτημα όπως αύριο μας κοινοποιήσετε τον κατάλογο των όσων υπέβαλαν αίτημα για ομιλία ενός λεπτού με δύο κριτήρια. Ότι δεν ομίλησαν στην προηγούμενη Ολομέλεια και δεύτερο κριτήριο το χρόνο υποβολής του αιτήματο. Σέβομαι απολύτως και το πρόσωπό σας και το Προεδρείο αλλά νομίζω ότι δεν είναι privilegium του Προεδρείου να κατανέμει το ρόλο κατά το δοκούν. Υπάρχουν ορισμένες αρχές και πρώτη αρχή είναι η αρχή της διαφανείας. Περιμένουμε αύριο να μας στείλετε τον κατάλογο και βλέπω ότι συμφωνούν και άλλοι και επιδοκιμάζουν και άλλοι συνάδελφοι με δύο κριτήρια όπως επαναλαμβάνω. Το κριτήριο του χρόνου υποβολής του αιτήματο και το κριτήριο το αν ομίλησα στην προηγούμενη ολομέλεια ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το κριτήριο που χρησιμοποιούμε, όπως ξέρετε, είναι μια ισορροπημένη κατανομή τοποθετήσεων μεταξύ πολιτικών ομάδων ανάλογα με το μέγεθος των ομάδων και δίνουμε προτίμηση σε αυτούς που δεν ομίλησαν στην προηγούμενη Ολομέλεια. Αυτά είναι τα κριτήρια που ακολουθούμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν μίλησε σήμερα ούτε ένας από την ομάδα των πράσινων ενώ από άλλες ομάδες μίλησαν και πέντε και εφτά άτομα. σας παρακαλώ. Μα αυτό εξήγησα αγαπητέ συνάδελφε προηγουμένως. Τρεις ζήτησαν το λόγο από την ομάδα σας. Και οι τρεις που είχαν ζητήσει το λόγο είχαν μιλήσει στην προηγούμενη Ολομέλεια. Οπότε εφαρμόσαμε αυτό το κριτήριο για να μοιράσουμε τις τοποθετήσεις ισορροπημένα. Ωραία. Να συνεχίσουμε τότε. Επόμενο σημείο. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, ποιος θα διαλέγει τα κριτήρια εσείς, οι υπηρεσίες, είναι γραμμένα πουθενά. Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Λοιπόν, έχουμε έναν κατάλογο με τους βουλευτές που ζήτησαν το λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 150. Και έχουμε τον κατάλογο όσων μίλησαν στην προηγούμενη Ολομέλεια. Και έτσι λοιπόν, όπως θα διαπιστώσατε, έδωσα το λόγο σε όλους τους ομάδες ε τώρα η τύχη το έφερε. Οι ομιλητέ των Πρασίνων να έχουν μιλήσει στην προηγούμενη Ολομέλεια, γι' αυτό δεν του προτιμήσαμε. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή, φροντίζουμε ο καθένας να μπορεί να μιλάει ανάλογα με τη βαρύτητα της ομάδας του και αν δεν έχει φυσικά μιλήσει στην προηγούμενη Ολομέλεια. Πολύ λογικό μου φαίνεται. Αλλά αυτό δεν είναι γραμμένο πουθενά σε κανέναν κανονισμό. Ούτε στον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Η Προεδρία με τις αρμοδιότητες που έχει διαλέγει τον τρόπο της πορείας της Ολομέλειας με δικαιοσύνη για όλες τις ομάδες. Κύριε Πρόεδρε, Μπορείτε να μου πείτε αν βρίσκομαι στον κατάλογο όσων ζήτησαν να παρέμβουν για σήμερα και αν είμαι στον κατάλογο όσων μίλησαν στην περασμένη Ολομέλεια. Τώρα μπορείτε να μου απαντήσετε. Να σας το πω αμέσως. Είστε η κυρία Παλιαδέλη. Είστε στη λίστα της σοσιαλιστικής ομάδας. η σειρά που δίνει το λόγο είναι αναλόγως με τη σειρά που έχει ε, ζητηθεί και έχει καταγραφεί. Οπότε δώσαμε το λόγο σε έξι ε, ευρωβουλευτές της πολιτικής σας ομάδας. Εσείς ε, και εσείς είσαστε στην χρονολογικά χρονολογικά σας λέγω δηλαδή από πλευράς χρονολογικής σειράς εσείς είχατε τον αριθμό 9 Εάν λοιπόν μου επιτρέπετε, ε, θα ήθελα να συνεχίσω τη συνεδρίαση. Σας εξήγησα ποια είναι τα κριτήρια. Τι άλλο θέλετε. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι καλό είναι να ξέρουμε εκ των προτέρων ποιος θα πάρει το λόγο. Είναι 10 η ώρα το βράδυ και καθόμαστε εδώ χωρίς λόγο, δεν παίρνουμε το λόγο. Θα πρέπει να έχουμε ένα κανόνα δύο ώρες πριν να γνωρίζουμε ποιος θα λάβει το λόγο για αυτές τις ομιλίες ενός λεπτού. Πρόεδρος, πολύ ωραία, θα λάβουμε υπόψη το έτοιμά σας. Πρόεδρε, δεν είναι δικό σας λάθος, αλλά είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Περιμέναμε ώρες εδώ για να πάρουμε το λόγο. Είναι 10 η ώρα και μας δίνουν χρόνο ενός λεπτού, αλλά δεν μπορούμε να ξοδεύουμε εδώ τον χρόνο για σημαντικά θέματα των περιοχών μας. Θα πρέπει να έχουμε το λόγο το, για να μιλήσουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε σε αυτό το κοινοβούλιο ότι εφόσον είμαστε εδώ θα πάρουμε το λόγο Καθόμαστε εδώ και περιμένουμε, αλλά οι πολίτες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι, έχουν βαρεθεί γιατί, με αυτά που συμβαίνουν εδώ γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικαιώματά τους. Οπότε τα έχουμε πει και στον κύριο Μπαρόζο, όλα αυτά είναι μια φάρσα. Είμαι εδώ 10 η ώρα το βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη τουλάχιστον θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε το λόγο για σημαντικά θέματα του κράτους μελουζά. Παρακαλώ, δώστε τα τώρα στους προϊταζεταμένους σας γιατί αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι δικτατορία. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μπαρόζο είναι πρόεδρος της Κομισιόν, όχι του Ευρωκοινοβουλίου. Λοιπόν, αν, αν δεν κάναμε όλε τούτε τι πλιαρίες και μπορούσαμε να τοποθετηθούμε ο, κανένα, ο καθένας από εμά, αντί να χρονοτριβούμε, επειδή είναι 10 η ώρα, ε, θα είχε πει ο καθένα το δικό του ερχόμαστε εδώ για να εκφράσουμε τους ε, εκλογείς μας. Λοιπόν, πραγματικά το βρίσκω αλαζονικό μετά να μας κόβουν και από τη λίστα. Λοιπόν, η κατάσταση είναι σαφέστατη. Εμείς έχουμε μισή ώρα για αυτόν το γύρο του ενός λεπτού. Εσείς ζητήσατε το λόγο πολύ περισσότεροι από όσοι γεμίζανε μισή ώρα. Και αυτό το οποίο κάνει η Προεδρία είναι να εφαρμόζει λογικά και δίκαια μέτρα σύμφωνα με τις εξουσίες που έχει. Καταλαβαίνω το πρόβλημά σας. Λοιπόν, με τον Διευθυντή των Υπηρεσιών της Ολομελίας θα μελετήσουμε μία φόρμουλα ούτως ώστε να έχουμε μία ιδέα πάνω κάτω γιατί ποτέ δεν θα είναι ακριβής για το πόσοι θα τοποθετηθείτε ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των όσων βρίσκονται σε αναμονή. Λοιπόν τώρα αν μου επιτρέπετε να συνεχίσουμε την Ολομέλεια διότι αλλιώ θα μείνουμε όλη τη νύχτα συζητώντα τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο σημείο τη σημερινής διάταξη. Φυσική καταστροφή στη Μαδέρα. Θεομηνία στη Μαδέρα. Εξ ονόματος της Κομισιόν, ο κύριος Σέτιγκερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές,